χωρίς να ζητήσει κάποιες τροποποίησεις. Ελπίζω ωστόσο αυτές να μπορέσουν να γίνουν μέσα σε ένα πνεύμα επικοδομητικής συνεργασία τις επόμενες εβδομάδες. Σας ευχαριστώ κύριε Σβάπ. Μάλλον πρόκειται να ξενυχτήσουμε, σας προεδοποιώ. Λοιπόν, κλείνει εδώ η συζήτηση. Αύριο στις 11.30 θα ψηφίσουμε. Επόμενο θέμα, προφορική ερώτηση προς την για την εφαρμογή της οδηγίας σε σχέση με την πέτα των καυσίμων. Ο συντάκτης, ή μάλλον η συντάκτρια της ερώτησης αυτής έχει το λόγο, η κυρία Μακάβαν. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κατάρχας. θέλω να ευχαριστήσω τη διάσκεψη των Προέδρων που βρήκε χρόνο να μπει αυτό το θέμα στη μέση διάταξη και ευχαριστώ και την Επίτροπο που βρίσκεται εδώ τόσο αργά. Είναι ένα θέμα ε, σημαντικό για το Κοινοβούλιο. Φαίνεται να είναι τεχνικό εκ πρώτης όψεως, γιατί αφορά τα μέτρα εφαρμογής ε, για την ε, οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων σε ό,τι αφορά ε, τη μέσα αναφοράς για τις εκπομπές καυσαερίων. Αλλά το σημαντικό θέμα και το σημαντικό μεγαλύτερο, το σοβαρότερο αν θέλετε, είναι πόσο σοβαροί είμαστε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των εκπομπών των συγκοινωνιών. Ξέρουμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό των εκπομπών προέρχεται από τα καυσαέρια και αυξάνεται το ποσοστό αυτό. Επομένως θέλουμε να είναι καθαρά τα καύσιμα των μεταφορών για να καταπολεμηθούν και κλιματικές αλλαγέ. Γι' αυτό και η οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων είναι σημαντική. Τώρα έχουμε αυτό το θέμα με την ασφαλτούχο άμμο, με το σχιστόλιθο που έχει πετρέλαιο. Υπάρχουν ε, κάποιες προτάσεις, οδηγίες έγιναν στο τέλος του χρόνου ε, υπήρξε κάποια καθυστέρηση όμως και γνωρίζουμε ότι στόχος, ε, μάλλον λόγος ήταν εσωτερική συζήτηση στην Κομισιόν για το κατά πόσο θα πρέπει σε αυτές τις ασφαλτούχες άμμους να δοθεί μια τιμή, μια βασική τιμή αναφοράς. Και μας είπαν ότι δεν μπορούμε να έχουμε μέτρα γιατί ε, οι μετρήσεις, γιατί δεν υπήρχε επιστημονική μελέτη που να τι προτάσεις της Κομισιόν πάντω ένα προώρο σχέδιο τη Κομισιόν. Είδαμε ότι υπήρχε μια τιμή ξεχωριστή ε, στο ε, πρώτο σχέδιο για τι ασφαλτούχες άμμους, αλλά αυτό τελικά ε, διαγράφηκε αυτό το όριο. Λοιπόν, τώρα έχουμε μελέτη, κυρία Επίτροπε, έχουμε μελέτη για τι άμμους, τις ασφαλτούχους και η μελέτη αυτή, η οποία δημοσιεύτηκε πριν από δύο μήνε δείχνει κάτι που κι άλλες μελέτες είχαν ήδη δείξει, δηλαδή ότι από καναδικές Ε, άμμους έχουμε πολύ σημαντικά ποσοστά σε σχέση με το συμβατικό καύσιμο και για το πετρέλαιο αποσχιστόλιθο 132-139 ε, ανά μεγατζούλιν εκπομπές του άνθρακα και στην πρώτη περίπτωση πάνω από 100 σε σχέση με το 81. Λοιπόν, άρα είναι πιο, ε, μεγάλη μόλις που εκπομπές καυσέρι που προέρχονται. Προτείνουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί αυτό υπόψη κατά την εφαρμογή τη οδηγία για την πέτα των καυσίμων. Δεν είναι όμω τεχνικό μόνο το ζήτημα. Την προηγούμενη εβδομάδα πολλοί βουλευτέ είχαν λάβει ε, μια αίτηση από χιλιάδε συμπολίτε μα οι οποίοι ανησυχούν για το θέμα αυτό. Θέλουν το ίδιο με αυτό που θέλω και εγώ. Δηλαδή μία ξεκάθαρη και σωστή επισήμανση στις ετικέτες για, αυτά τα, για τις ασφαλτούχες άμμους. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Στην Καλιφόρνια ήδη υπάρχει ένα ειδικό πρότυπο ε, και θεωρούνται ότι οι ασφαλτούχες ε, άμμοι περιέχουν πολύ μεγάλα ε, ποσοστά άνθρακα, δεξιδίου του άνθρακα. Έχουμε τα λόμπι που ασκούν πιέσεις και ξέρουμε ότι ακόμη και τώρα που γνωρίζουμε ότι αυτά τα πετρώματα είναι πιο ε, ρηπογόνα σε σχέση με το συμβατικό καύσιμο, λένε α κερδίσουμε λίγο χρόνο ακόμη να κάνουμε κάποιε μελέτε. Όμω ε, δεν συμφωνώ, δεν νομίζω ότι πρέπει να ε, καθυστερήσουμε, γιατί η ασφαλτούχια άμυ είναι μια, ένα από τα πιο ρηπογόνα ε, μέσα για να έχουμε καύσιμο των μεταφορών. Θα πρέπει να δούμε πώς θα κατηγοριοποιηθούν οι άμοι αυτοί στην ε, οδηγία γιατί αλλιώς ε, τα κάψιμα των μεταφορών θα γίνονται όλο και πιο ε, βρώμικα αντί να γίνονται πιο καθαρά. Θα δούμε σε λίγο πόσοι από τους συναδέλφους θα συμφωνήσουμε με τις δικές μας ανησυχίες. Γνωρίζουμε εσείς πόσο, κύριε Επίτροπε, είσαστε ευαισθητοποιημένοι σε αυτά τα θέματα της κλιματικής αλλαγής και ελπίζουμε ο δικός χάρτης για μικρή μικρής σε άνθρακα καύσιμα ε, θα το περάσετε αυτό. Ελπίζω να μας δώσετε κάποια καλά νέα κύριε Επίτροπε και να μας πείτε τις επόμενες εβδομάδες θα έχετε τα πρότυπα εφαρμογή και θα έχουμε υψηλή τιμή για το σχιστόλιθο που παρέχει πετρέλαιο και για τι ασφαλτούχε άμμου. Σα ευχαριστώ κυρία Μακάβαν. Το λόγο έχει η Επίτροπο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως ακούσαμε από τη Λίντα Μαγκάβαν, συμμεριζόμεθα την άποψη στην Επιτροπή για το πόσο είναι σοβαρό να αντιμετωπιστούν τα θέματα των εκπομπών στις μεταφορές και αυτό φαίνεται και στις προτάσεις που κάναμε σήμερα για τις μεταφορές οι εφαρμοστικές διατάξεις σε σχέση με τους στόχους περιορισμού της εκπομπής διοξιδίου του άνθρακα είναι κάτι το οποίο πάντα λαμβάνουμε υπόψη μας. Η καθυστέρηση όμως δεν θα μειώσει την ικανότητά μας να πετύχουμε τους στόχους μας γιατί καμία χώρα δεν έχει θέσει ενδιάμεσους στόχους για το 2014. Προετοιμάζοντας την πρότασή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει υπόψη ότι οι ρυθμίσεις θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους το περίπλοκο και ε, γενικά το ευαίσθητο θέμα της συλλογή χαρακτηριστικών για τα διαφορετικά καύσιμα. Στις, το προηγούμενο φθινόπωρο και στις αρχές του 2011 έγιναν συζητήσεις ε, στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, παίρνουν τώρα την τελική μορφή τους και θα υπάρξουν κάποιες συζητήσεις τους επόμενους μήνες. Σχετικά τώρα με τις ε, ασφαλτούχες άμμους και τους, ε, και τους χιστόλιθους που παράγουν πετρέλαιο, είναι σαφές ότι τα επίπεδα ε, μόλυνσης δεν είναι ακόμα απόλυτα δεδομένα. Τώρα έχουν υπάρξει βέβαια συγκεκριμένες εκθέσεις οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι εκθέσεις αυτές θα πρέπει να περάσουν μέσα από μια διαδικασία ελέγχου αξιοπιστίας. Έχω έρθει σε επαφή ε, με τους υπεύθυνους συναδέλφους επιτρόπους ε, που ασχολούνται με τα θέματα του εμπορίου έτσι ώστε η στάση μας ε, να είναι συμβατή με τις υποχρεώσεις που έχουμε σε σχέση με το παγκόσμιο εμπόριο. Χωρίς να θέλω λοιπόν να προκαταλάβω τις περαιτέρω διαβουλεύσεις και τις τελικές αποφάσεις, είναι πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αυτή τη φάση να προτείνει κάποιες πρώτες εφαρμοστικές διατάξεις στην Διακανονιστική Επιτροπή, η οποία θα λάβει υπόψη τις συγκεκριμένες προτάσεις επιπέδων μόλυνσης για την άμμο και τα, τους χιστολίθους, όπως επίσης και για τη μετατροπή φυσικού αερίου σε υγρά Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θα μελετήσει επίσης ε, και τις ε, δυνατότητες για την πιθανή δημιουργία των ενεργειακών χαρακτηριστικών ορισμένων ζωοτροφών. Η διαδικασία για τη διαμόρφωση των νέων κατηγοριών έχει ξεκινήσει. Εξετάζουμε τις νέες αυτές προτινόμενες κατηγορίες και θα καταλήξουμε σε ένα κατάλογο όταν έχουμε συλλέξει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία. Συνεπώς, Πρόεδρε, μιας και χρειάζονται κάποιες εβδομάδες για, την, για τον έλεγχο αξιοπιστίας των εκθέσεων αυτών, θα υπάρξει μια κάποια καθυστέρηση πριν από τις πρώτες εφαρμοστικές διατάξεις συνολικά για το πακέτο αυτό όταν έχουμε τα στοιχεία και όταν γίνουν δεκτά από την, από την αρμόδια ρυθμιστική επιτροπή, τα αποτελέσματα θα σας έλθουν για εξέταση. Ευχαριστώ Επίτροπε. Περνάμε στους ομιλητές εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων. Για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, δύο λεπτά, ο κύριος Σνέλχαρτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ την κυρία Μακάβαν για την κατάθεση της ερωτήσεως διότι με την οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων επιβάλλεται η μείωση των ε, εκπομπών οξυδίων του άνθρακος σε όλο τον κύκλο ζωής του καυσίμου από το δηληστήριο μέχρι την καύση του από το 2011 οι εκπομπές αναμονάδα ε, καυσίμου θα πρέπει να έχουν μειωθεί μέχρι το 2020 κατά 10%. Αυτό θα είναι δυνατόν μόνο εάν υπάρχουν στάνταρτ τιμές, οι οποίες τιμές πρέπει πλέον να θεσπιστούν και να οριστούν. Θα ήθελα και το είδα και με την κατάθεση της ερωτήσεως της κυρίας Μακάβαν ότι κάπως θέλει να βγάλει απ' έξω από την παραγωγή ορισμένους τύπους καυσίμων. Εδώ όμως χρειάζεται προσοχή, διότι υπάρχουν διαφορετικές έρευνες σχετικά με το πετρέλαιο που βγαίνει από άμμο ή από σχιστολίθους. Μίλησα πριν από λίγο με έναν εκπρόσωπο της βιομηχανίας αυτής που μου λέει ότι υπάρχει σημαντική εξέλιξη που μπορεί να οδηγήσει σε πολύ καλύτερη εξέλιξη, σε πολύ καλύτερη ε, απόδοση. Και μην λησμονούμε ότι υπάρχουν και ενεργειακέ πηγέ εκτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και τον πόρο αυτό τον διαθέτουμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα θα πρέπει να περιληφθεί και αυτή η διάσταση στην συζήτηση. Βέβαια, όλα αυτά θα προχωρήσουν όταν υπάρχουν πρώτα οι απαραίτητε τιμέ, όταν θεσπιστούν δηλαδή και γίνουν γνωστέ οι τιμέ. Σα ευχαριστώ κύριε Σνερχάρτ. Εξ ονόματο των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, για δύο λεπτά ο κύριος Αρσένης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ε, επίτροπε, συνάδελφοι. Πραγματικά ήταν ένα πάρα πολύ κρίσιμο ζήτημα. Είναι τρεις με πέντε φορές περισσότερες εκπομπές ε, από την παραγωγή πετρελαίου από Τάρσανς, από Μόδι Πίσα, σε σχέση με άλλες μεθόδους παραγωγής. Και αυτός ο πολυπόθητος δείχτης που θέλουμε να υπάρξει μέσα στην οδηγία θα μας ε, επιτρέψει να μην επιδοτήσουμε αυτή την καταστροφική μέθοδο παραγωγής. Είπατε ότι ε, έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και όμως παρόλα αυτά που έχουμε μελέτη, παρόλα αυτά που αυτό είχαμε πει, ότι μας λείπει μόνο η μελέτη για να προχωρήσουμε. Θέλουμε τώρα αυτή η μελέτη να έχει περάσει από, ένα, από peer review. Το ερώτημα είναι, ε, Επίτροπε, πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία ποια είναι τα χρονοδιαγράμματα πόσο ακόμη θα περιμένουμε μέχρι αυτός ο δείκτης να είναι ελεγμένος και μέσα από αυτή τη μεθοδολογία και επιτέλους να μπορέσουμε να τον βάλουμε στην ομοθεσία μας. Γιατί πραγματικά δεν είναι μόνο οι εκπομπές το πρόβλημα με την αμμοδιπίσα. Είναι και η καταστροφή ε, μοναδικών δασών κρίσιμων συμμάχων μας για την αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής των Boreal δασών της, ε, του Καναδά. Την ίδια στιγμή καταστρέφουμε τη γη των Ιθαγενών στην οποία γίνεται αυτή η τεράστια καταστροφή και αν δεν βάλουμε το δίχτυ στην νομοθεσία μας σήμερα ε, αυτή η καταστροφή θα εξαπλωθεί και σε άλλες χώρες. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κυρία Αρσένη για τους ε, φιλεύθερους δημοκράτες. Κυρία Χόλ για δύο λεπτά. Θέλω να ευχαριστήσω την Επίτροπο Κάρτ κύριε Πρόεδρε, για τι μακροχρόνιες προσπάθειέ τη και για τη θετική ανακοίνωση την οποία προέβη σήμερα το βράδυ. Έχετε συναντήσει πολλέ φορέ ευρωβουλευτέ και σίγουρα δεν οφείλεται σε εσά ε, το πρόβλημα ε, και η εμπλοκή που παρουσιάστηκε. Πάντω είναι όλα πολύ απογοητευτικά. Αρχικά φάνηκε δεν αρκούν πια όλες αυτές οι μελέτες που δείχνουν ότι είναι πολύ μεγαλύτερη εκπομπή ε, αερίων ε, ρηπογόνων σε σχέση με το ρηπογόνο καύσιμο και ότι έπρεπε να γίνει μία έρευνα, να έγινε λοιπόν και από το Κοινό Κέντρο Ερευνών που δείχνει ότι έχουμε αύξηση σε σχέση με το 51% ε, του σημαντικού κασίμου. Τώρα λέτε δεν αρκεί αυτό, θέλουμε peer review. Δεν χάνουμε έτσι χρόνο. Και κρίμα είναι το ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλη πίεση από τους λομπίστες για την αμμοδιπίσα. Γιατί εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε κάποιες διακρίσεις και συγκεκριμένα κατά του Καναδά. Γιατί υπάρχουν και πολλοί άλλοι χώροι στη, ε, για αμμοδιπίσα, όπως και, στο Ηνωμένο, και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα είναι ότι υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον σε παγκόσμιο επίπεδο ε, για την παραγωγή πετρελαίου. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει και να επιμείνουμε ξεχωριστή τιμή. Γιατί αλλιώ η αμμόδη πίσα θα παίρνει όλο και μεγαλύτερο μερίδιο στο ενεργειακό μείγμα. Και ίσω φτάσουμε σε μια κατάσταση όπου τελικά θα έχουμε του στόχου μα του 6% μείωση, όπω προβλέπονται από τι οδηγίε, στο χαρτί, αλλά στην πράξη θα έχουμε υψηλότερε εκπομπέ από τη σήμερα. Θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο να εξηγήσετε στη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Τρέιντ, όπως φαντάζομαι ότι έχετε κάνει, ότι δεν θέλουμε να επιτεθούμε στον Καναδά. Σε καμία περίπτωση το Κοινοβούλιο θέλει να υπάρξουν αυτές οι τιμές, θέλει να λυθεί το όλο ζήτημα για να υπάρξει μια ομαλή μετάβαση και σε σχέση με την εμπορική συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Καναδά. Σα ευχαριστώ κυρία Χολ. Μέρος των Πρασίνων, κυρία χάσει για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Υποτίθεται ότι θέλουμε να μειώσουμε κατά 6% τις εκπομπές. Μα θα ήταν παράλογο να πάρουμε αυτές, αυτά τα πιο ε, ρηπογόνα καύσιμα τα οποία, των οποίων εξόριξη γίνεται και στον Καναδά αλλά και στην Αφρική και αλλού. Πρέπει να δούμε λίγο σοβαρότερα το θέμα. Η κυβέρνηση του Καναδά ασκεί πίεση λόμπι. Αυτό δεν είναι παραδεκτό. Εάν έχουν, αν πιστεύουν άλλα πράγματα στον Καναδά, θα πρέπει να αποδείξουν την ισχύ των επιχειρημάτων τους. Τα ίδια λέμε εμείς και για τα βιολογικά καύσιμα που πρέπει η σύγκριση της αξίας τους να γίνει και με άλλους πόρους ενέργειας. Ο κύριος Σόνικ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Υπάρχουν ε, πάρα πολλές περιοχές ε, με ασφαλτούχες άμμους. Πολλοί θεωρούν ότι θα μπορούσαμε να παράγουμε καύσιμα από εκεί σε διπλάσια ποσότητα από ό,τι μπορούμε να κάνουμε ε, με την παραδοσιακή μορφή εκμετάλλευσης του πετρελαίου. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με μία σύγκρουση από τη μία μεγάλη ανάγκη νέους πόρους για νέους ενεργειακούς πόρους και από την άλλη προβλήματα σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, των δασών και του υδάτινου ορίζοντα. Θα πρέπει να πιέσουμε τις επιχειρήσεις οι οποίες εμπλέκονται στη δραστηριότητα αυτή να φυτεύουν νέα δέντρα στις περιοχές τις οποίες εκκερσώνουν ένα τμήμα των κερδών θα πρέπει να απευθύνεται στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να στηρίξει τις τεχνολογίες οι οποίες μειώνουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Καναδάς είναι διασυνδεδεμένοι οικονομικά, υπάρχει ταύτιση συμφερόντων και βιομηχανικών, όχι μόνο οικονομικών και γι' αυτό ακριβώς και οι καναδικές επιχειρήσεις θα πρέπει να συμπεριφέρονται ανάλογα με τις ευρωπαϊκές ρυθμίσεις και κανόνες. Ευχαριστώ κύριε Σόνικ. Λίζα. Ευχαριστώ. <clears throat> ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι. Πρώτα ευχαριστώ την Λίντα Μακάβαν που ανέλαβε την πρωτοβουλία. Ευχαριστώ και την πίτροπο Κόνι Χέντεγκάρντ που ανταποκρίθηκε δεν μας ικανοποιεί βέβαια η ταχύτητα, αλλά γνωρίζουμε ότι βρίσκεται σε καλά χέρια το θέμα, στα χέρια της κυρίας Σέντεγκάρτ. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν συζητήσεις και εντός της Κομισιόν, αλλά και με άλλους ενδιαφερομένους φορείς. Είναι γεγονός ότι η αμμώδης πίσα έχει σημαντικές οικολογικές συνέπειες. Ίσως αμφισβητούνται κάποια νούμερα, αλλά το γεγονός ότι υπάρχει τεράστιο οικολογικό πρόβλημα νομίζω δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Όταν συζητούμε εντατικά για τις επιπτώσεις που έχουν τα βιολογικά καύσιμα, μέχρι και να συζητούμε για ενδεχόμενη μείωση παραγωγής τροφίμων λόγω της παραγωγής καυσίμων, θεωρούμε, ε, αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντική είναι η ε, πρωτοβουλία της κ. Μακάβαν. Όπως λέει και ο υπουργό Περιβάλλοντος στη Γερμανία, ο Νόρμπερτ Ρέτκεν, έχουμε ήδη πάρει τα εύκολα, τα όρημα φρούτα που ήταν πιο χαμηλά που πρόσφεραν τα ορυκτά καύσιμα. Τα έχουμε ήδη συλλέξει αυτά. Τώρα γίνονται πιο δύσκολα τα πράγματα. Όλοι έχουμε λοιπόν λόγο και μάλιστα και με τα πιο πρόσφατα γεγονότα των τελευταίων ημερών να επανεγκύψουμε στο θέμα της απόδοσης της ενέργειας, της αποδοτικής χρήσης της ενέργειας, να επιμείνουμε στην προσπάθεια επίτευξης του στόχου της μείωσης 20%, να ακούσουμε και από τον Επίτροπο που είναι αρμόδιος για τις μεταφορές, αλλά όχι λόγια, να δούμε συγκεκριμένες προτάσεις και αυτές να έρθουν τώρα και όχι στην επόμενη περίοδο. Σας ευχαριστούμε κύριε Λύση. Περνάμε στη διαδικασία Catch the Eye. Ο κύριος Γκέρ Μπράνι για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Γίνεται εδώ μια έκθεση φωτογραφίας για τις αμμώδεις πίσες στον Καναδά. Βλέπει κανείς φωτογραφίες υπέροχων δασών και μετά υπάρχει ένα χάσμα και βλέπει κανείς τεράστιους λεκέδες πετρελαίου σε τεράστιες εκτάσεις. Αξίζει να πάει να δει κανείς αυτή την έκθεση. Εκτός από την τεράστια απώλεια βιοπικιλότητας, όλη αυτή η υπόθεση έχει και σημαντικές εκπομπές διοξιδίων του άνθρακα. Αυτά για μένα είναι λόγος αρκετός για να αντιταχθώ στην εξόριξη πετρελαίου από τις αμμώδεις πίσες του Καναδά. Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να περιλάβουμε τις σχετικές τιμές στην οδηγία ποιότητας των καυσίμων. Άκουσα τα όσα είπε η κυρία Χέντεγκαρτ και υποθέτω ότι θα το πράξει. Ελπίζω ωστόσο να αντιταχθεί στην περαιτέρω εξόριξη ε, πετρελαίου από αμμώδεις πίσω στον Καναδά. Ευχαριστώ για ένα λεπτό κυρία Τικάου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε για να μειωθεί κατά 20%, για να μειωθούν μάλλον ε, οι εκπομπές κυπριακών αερίων μέχρι το 2020, πρέπει να έχουμε σημαντικά αποτελέσματα και να επενδύσουμε σε μέτρα για την μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση του τομέα τη οικοδομή και του τομέα των μεταφορών. Όταν εγκρίναμε την οδηγία για την ε, ποιότητα των ε, καυσίμων για τον τομέα των μεταφορών έγιναν πολλέ συζητήσει ο κλάδος της τότε είχε θεωρήσει ότι χρειάζεται μια πιο μεγάλη χρονική περίοδος για να αυξηθεί το ποσοστό των βιοκαυσίμων. Για να δούμε ποια είναι η πίωση ατμού που μπορεί να ε, δεχθεί το όχημα κτλ. Και, και να υπάρξουν τα σχετικά πρότυπα. Πρέπει να γίνουν λοιπόν επενδύσεις και στον τομέα της εκπομπή ρηπογόνων, ε, ε, ρήπων για τι επογόνε εκπομπέ. Για να ελέγξουμε και να μειώσουμε τι εκπομπέ από το μέτρο μεταφορών θα πρέπει να επενδύσουμε κυρίω στην ανάπτυξη ενό εφιούς ηλεκτρικού δικτύου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο θα είναι σε θέση να συμπεριλάβει και τι τοπικά παραγόμενε ενέργειες, μιλώ για τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, αλλά και για τα ηλεκτροκίνητα οχήματα. Σα ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Μέσαρος για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, πρέπει να πω ότι οδηγεί αυτή μάλλον θα καθησυχάσει τα δηληστήρια χωρίς να έχει τεθεί βέβαια ακόμη σε ισχύ. Ε, θέλουμε να δούμε ακριβώς ε, πώς θα μετρώνται εκπομπές, αν θα υπάρχει μια σταθερή μέθοδος, αν θα έχουμε ένα μέσο όρο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αν θα έχουμε μια υβριδική μέθοδο που είναι μια εναλλακτική μορφή υπολογισμού. Οι εκπομπές θερμοκυπριακών αερίων θα πρέπει να μειωθούν. Και έχουμε στείλει μια επιστολή στην Επίτροπο. Μας απάντησε η Επίτροπος, μεν, αλλά δεν απαντάει και στα ερωτήματα η επιστολή. Δεν καθισχάσει τι ανησυχίες μας δεν πρέπει να τεθούν ε, τα δηληστήρια σε ανταγωνιστικό μειονέκτημα υπέρ του ρωσικού πετρελαίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μέσαρος. Για ένα λεπτό κύριο Σκέλη. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι Θα ήθελα να ήμουν μέλος της Επιτροπής. αν κάποιος λοιπόν φύγει από εσά θα ήθελα να έλθω εγώ. Τέλος πάντων, εννοώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χρειάζεται να γίνει περισσότερη δουλειά για τα κτίρια, για τις μεταφορές. Σε ό,τι αφορά τις ίδιες μεταφορές, νομίζω ότι χρειάζεται να γίνει πολυ πολύ περισσότερα πράγματα. Πρώτα-πρώτα στην παραγωγή αυτοκινήτων, στην αυτοκινητοβιομηχανία, να φτιάξει αυτοκίνητα που να παράγουν λιγότερους ρήπους. Σχετικά με το εδώ το θέμα, εμείς ως αντιπροσωπεία κάναμε μια σχετική επίσκεψη, μας έδειξαν και τις τεχνολογίες που αναπτύσσονται και θα πρέπει να έχουμε ανοιχτό μυαλό απέναντι στην εκμετάλλευση του πετρελαίου από τους σχιστολίθους και άμμους. Ευχαριστώ. Ναι, κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο για το πολύ ξεκάθαρο μήνυμα που δώσατε απόψε. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο. Και πράγματι υπάρχει αυτή και η αίσθηση ότι ήταν επίγον, γι' αυτό και υπήρξαν υπόμονο το Κοινοβούλιο και ο κύριος Αρσένης που μιλήσαν για το χρονοδιάγραμμα, πότε θα τελειώσει όλο αυτό. Πρέπει να σας πω ότι μιλάμε για ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Μιλάμε για αυτό το peer review κάποιες εβδομάδες και μετά θα πρέπει να επανέλθει αυτή η εξολόγηση στην Κομισιόν, να έχουμε την εσωτερική μας διαδικασία και στη συνέχεια θα περάσουμε στην επόμενη φάση, δηλαδή ε, κράτη-μέλη. Κοντεύουμε δηλαδή. Όπως έλεγε η κυρία Χολ, το θέμα δεν είναι να πάρουμε πρωτοβουλίες που θα συνιστούν ε, διακρίσεις και όλοι καταλαβαίνουμε γιατί είναι σωστό να υπάρξει τεκμηρίωση και ε, ισχυρή έγκυρη τεκμηρίωση. Αυτό κάνουμε. Ξέρουμε ποιοι είναι οι λόγοι. Ένας από τους λόγους είναι και δεν συμπεριελήφθη ευθύ εξ αρχή όταν ξεκίνησε εδώ και χρόνια αυτή η υπόθεση. Τώρα όμω γίνεται αυτή η δουλειά και έτσι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε. Ολοκληρώνοντα, θέλω να πω ότι σε ό,τι αφορά για τις τιμές αυτές τις ε, ε, πίσες, η όλη καθυστέρηση για την υλοποίηση της οδηγίας, τι σημαίνει ουσιαστικά. Θα μπορούσαμε την τιμή αυτή, τη βασική την τιμή αναφοράς, να την έχουμε και να τη συμπεριλάβουμε ακριβώς στο ίδιο γύρο, στο, στο γύρο εφαρμογής της οδηγίας και να μπορούμε πιο γρήγορα πλέον να καθορίσουμε αυτή την τιμή για την αμμόδη πίσα. Αυτό δεν ήταν σίγουρο όταν ξεκινήσαμε πριν από 8 μήνες περίπου, 9. Σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ για όλους που εργάζεστε για να καταφέρουμε να φέρουμε σε αίσιο πέρας αυτή την υπόθεση. Σας ευχαριστούμε κυρία Επίτροπε. Περνάμε στο επόμενο σημείο της μερίσιας διάταξης, έκθεση κυρίου Σόλτς για τις γενικευμένες δασμολογικές προτιμήσεις. Πρώτος έχει το λόγο εισηγητής, ο κύριος Σόλτ.